Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα να αρχίσουμε. Μεταξύ άλλων, διότι έχουμε και πολλή δουλειά σήμερα και πάρα πολλές ψηφοφορίες. Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Και πριν τις ψηφοφορίες θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από την περιφέρειά μου και τους ευχαριστώ που ήρθανε. Τώρα τα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έχουν φτάσει. Σας ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, αρχίζουμε. Το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη που είναι εντολή για το τριμερή διάλογο 2016 προπολογισμό. Είναι η έκθεση ενός λαβία Λοιπόν, πάμε. Ψηφίζουμε. Η τροπολογία παρήθμων 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο. Σε τρία τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Το δεύτερο είμαστε. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρο, Είναι κρίση. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε δεν ξέρω αν ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται λοιπόν Πάμε στη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7. Σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά ελέγχομαι. Avete votato tutti? Ψηφίσαμε όλοι. στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Emendamento 10. Chi è a 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 σε 2 τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές ελέγχομαι Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Υπε, ε, δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές ελέγχομαι. Avete votato tutti? No, c'è un non iscritto di troppo. Υπάρχει μία εγγεγραμμένος. Έχει, πέρασε, έχει κλείσει η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, εγκρίνεται. Η συμβατική 2, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά το σχέδιο έτσι όπως έχει προκύψει με τις τροπολογίες. Παρακαλώ.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 το σημείο 10 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πρόκειται για την απόφαση έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων υπό το άρθρο 73 Food and Feed. Επίσημη έλεγχη. Παρακαλώ ψηφίζουμε.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 Votare il punto Θα ψηφίσουμε τώρα για το σημείο 11 αποτελεσματικότητα των πόρων και κυκλική οικονομία η κυρία Πιέτικα είναι η συγκήτρια. Θα πάμε αμέσως σε ψηφοφορία στην τροπολογία 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Όχι, στο συγγνώμη. Τροπολογία 78 της κυρίας Ντάλλη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 2 της ε, Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3 τμήμα 1 ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 82, 82 και 83 ταυτόσημες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. 84 έχει αποσυρθεί, 85 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 Μόλναρ υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική εξί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 της έμπλα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ναι, δεν είπα για αποχές, ζητώ συγγνώμη. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103. Όχι. Λέει ο Πρέπει να ψηφίσουμε την πάραφο 14 της ΕΜΠΛ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 της έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4 της έμπλ. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Λοιπόν, πέρα ψηφοφορίες και απορρίπτεται. Ε, 5 της έμπλα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 6 της έμπλα υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Πάφο 8 της έμπλα υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Πάω σε 9 της έμπη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι. Έλεγχος λέει τώρα ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Peras, Απορρίπτεται. Πάφος 10 έμπλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές εγώ θα έλεγα ότι εγκρίνεται αλλά το ελέγξουμε Avete votato tutti il voto è chiuso Εγκρίνεται. Εκατόν εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν έντεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εκατόν δώδεκα Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία μάλλον παράφος 18 έμπλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 και αφαβόρε. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά ελέγχουμε Avete votato tutti, il voto è chiuso. Οπωσδήποτε απορρίφθηκε. Λοιπόν, 177 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 183 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε εδώ. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Πέρας, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 194 και 195 Ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λοιπόν, τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την παράγραφο 6 της Ήτρε. Το πρώτο τμήμα. Without eco design κτλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα 215 του Τούρβε σε, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 219 ε, υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Peras απορρίπτεται. 2.21 υπέρ. κατά. Αποχέ. Δεν ξέρω τι κάνουν οι σιαλιστές τώρα εδώ. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, εκρίνεται. Δεν υπήρχε ούτε, ούτε χέρι δεν είδα. Τι να κάνω. Λοιπόν, 2.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.28 με μία προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογίες 2.34 και 2.35 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Πέρα aperifti, Απερίφθη. Απερίφθησαν. 14 τρίτο τμήμα τώρα Τη ΣΥΤΡΕ, Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti, il voto è Απορρίπτεται. 2.49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο έχει καταπίπτει 2.51 όχι η συμπαθική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 5 πρώτο τμήμα της ε, πρότασης Ήτρε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 πρώτο τμήμα της έμπλα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Adesso votiamo. Τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 13 δεύτερο τμήμα της Ήτρε υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Avete votato Ελπίζω να έχετε ψηφίσει όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 284 τούρμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 292 σε δύο τμήματα. Το πρώτο, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ...2.93... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... Votiamo adesso l'emendamento 296 e υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Απορρίπτεται. 297 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ψήφισε τροπολογία 299 ψήφι πε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 300 υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 303 υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 304 υπέ. κατά αποχές απορρίφθηκε. 305, υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να ψηφίσουμε και την παράγραφο 9 της Επιτροπής Ήτρε. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα ψάμε στην τροπολογία 305. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 306 είπε, Κατά. Αποχές έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική 21. ψηφίπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψήφι π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 15 της ίδιας Επιτροπής. Ψήφι π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Πρώτο τμήμα της ΣΥΤΡΕ. Ψήφι π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 της Επιτροπής Βιομηχανίας πάλι υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την παράγραφο 13, πρώτο τμήμα της Επιτροπής Ήτρα. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 14, το πρώτο τμήμα, τη ΣΥΤΡΕ πάντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 320, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 321 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 322. ψηφίπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 3, 29 και 30 μαζί. είπε. είναι ταυτόσιμες. Κατά αποχές απορρίφτονται. Παράγραφος 17 της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 335. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 336. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 337. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Η συμβαστική 25. Ψηφί Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο παράγραφος 8 της Επιτροπής Ήτρε. Ψηφί Κατά. Αποχές απορρίψεται. Τροπολογία 345. Ψηφί Κατά Αποχές. απορρίφτεται. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Δεν είδα καλά. Η 345 είπε, Εγκρίνεται. Η 72 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 346 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την 354 τώρα που είναι συμβατή με την 26 τη συμβαστική υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 359. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Περισσεύει ένα σοσιαλιστή και δημοκράτη. Ματίας, λέω, είστε υπεράριθμοι. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 362 και 473 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 363 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. 366 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 367 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 29 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 393 είπε. κατά αποχές απορρίψεται. Η τροπολογία 375 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 376 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 377 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψεται. Η τροπολογία 378 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 379 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίψετε. 380 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα μέσω πάμε στην τροπολογία 390. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 391 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 392 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 394 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 395 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 397 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε αμέσω στην 307, διότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της προηγούμενης, αφού το πρώτο απερίφθη. 307 ψήφι υπέρ. Κανείς δεν είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το τρίτο τμήμα της παραγράφου 13 της Επιτροπής Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18 Ήτρε ψηφί Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε την παράγραφο 19 της Επιτροπής Ήτρε υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Ψηφί Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Votiamo adesso. Τώρα θα ψηφίσουμε. Μισό λεπτό. Θέλετε παλήθευση του προηγουμένου. Πολύ ωραία. Ό,τι πείτε εσεί. Επαληθεύουμε τη συμβαστική 31 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα η παράγραφο 16 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 11. Όχι, 16 διορθώνει ο πρόεδρος της Ήτρε. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 11 τώρα Τη ΣΥΤΡΕ. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 12 της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 409. Ψηφί Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 410 Υπέ κατά, αποχές εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα τώρα της παραγράφου 20 της Επιτροπής Ήτρε, φυπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 11 της Επιτροπής Απασχόλησης, ψηφί Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 411 τροπολογία ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 7 της Επιτροπής Ήτρε ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 412 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 413 επέ κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 414 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 415 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τροπολογία 416 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 417. Νιπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Συμβιβαστική 32 τμήμα πρώτων. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 τμήμα δεύτερον. υπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 427. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το συμβασμό 33. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 437 ε, του συναδέλφου Λάινεν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 438. Ψήφι Κατά Αποχές απορρίπτεται. 439 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 444 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίψεται. Η τροπολόγια 445. Ψηφί περ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολόγια 446. Ψηφί περ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Ψήφι περ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την παράγραφο 7 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της παραγράφου 21 της Επιτροπής Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα τώρα, στην ίδια παράγραφο της Ήτρε, ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22, πάντα της Ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 ήτρε ψηφίπε κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 456. Ψηφίπε κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολόγια 457 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 459 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική υπαριθμό 36 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε την 467 τροπολογία τώρα Πε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 468 είπε. Κατά αποχές απορρίψεται. 469 και 470 είναι μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η τροπολογία 471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Η 472 υπέρ κατά έλεγχος. Sorry stop, stop. <laughs> Doesn't stop, stop. Okay. Now we can vote. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Votiamo il, eh, l'emendamento. Ε, 474. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 475. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 477 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 476. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ή 478 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε στις επόμενες τροπολογίες. Είναι υπαριθμόν 1 καπούτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 4, 5, 6 είναι ταυτόσιμες αυτές μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι 7 και 9 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Οι 10 και οι 55 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 11 και οι 12 είπε κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 24 και 25 που είναι ταυτόσιμες είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 25 τώρα είπε κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 2 Υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 Υπέ, ε, συγγνώμη Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 31 ε, Παουλούτσι Μποναφέ υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην 36. Ψηφί πέρα. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 37 και 38 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά απόχες ηλεκτρονική επαλήθευση Avete votato tutti? Eh, ψηφίσατε όλοι πέρα; Respinto. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 45-46 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47, 48 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Avete votato tutti, il voto è Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία που 49 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 ΠΕ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά απορρίπτεται. 53 υπέρ και κόντο κατά αποχές το ΕΛΚ τίποτα, υπέρ. Α, εγκρίνεται λοιπόν. Η τροπολογία 54, υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. Η 56, υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 57, υπέρ. Κατά. Απόχες, εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά το σύνολο όπως τροποποιήθηκε. Πολύ περίπλοκο κείμενο. <laughs> το κείμενο στο σύνολό του. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αντρέα. Κομπλιμέντια αλλά Χαρητήρια στην συγκήτρια. Πιετικάινεν. Ε, σας ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις ε, καθώς και όλους όσους σημαντικά συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση. Παρότι είχαμε σοβαρές διχογνωμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, θα αξίζουν ε, τα χειροκροτήματα και, τα, και οι ευχαριστίες ε, σε όλους. Σύρπα <laughs> πρέπει να μάθεις Ιταλικά, ειλικρινά. Okay. We can go to the next. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο σημείο της διάταξη σε ψηφοφορή για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ελεονόρα Εύη είναι η συγγήτρια. Αν είστε έτοιμοι, να αρχίσουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 50 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 51 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 επτά της ε, Γκαρσία Πέρες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά Απόχες εγκρίνεται. Τώρα. 86, Λουζί και Μίλλερ, υπέρ. Κάτα. Απόχες. Ελκ. Υπέρ είσαστε. Ωραία. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. κατά απόχες εγκρίνεται Αστική 6 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται. 109 υπέρ κατά αποχές ένα μία επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε πέρας, εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά Απόχε. εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά Απόχε. εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, έρχεται. Il voto è chiuso. Πέρας, εγκρίθηκε. Now we can vote the behind. Τώρα σημείο 13. Λίνσα για τις ε, ε, ζωοτροφές. Μπορούμε να αρχίσουμε, άμα είσαστε έτοιμοι. 19. Α, ε, μπλοκ. Μου. 19, 76, 77, 220, 221, 222, 24, 30 και 38. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 156. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157, 158, 18 και 111 μπλοκ παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τώρα μπλοκ πάλι. 20, 159, 112 και 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτονται. Η συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Το δεύτερο τμήμα της 84 της συναντέλφου Μίλλερ είναι προσθήκη. Υπέρ. Α, ναι, με την προφορική τροπολογία που ζήτησαν οι φιλελεύθεροι. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για την προφορική. Όχι. Τότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τώρα τις ε, ταυτόσιμες 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αμπλοκ 88 και 94 μαζί παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 97-98 είναι ταυτόσημες μαζί παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 99 και 100 ταυτόσιμες επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται unblock τώρα 89 και 90 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται 8 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εννέα. Οι σε 9, 105 και 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 10, 107, 108 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 11, 109, 110 είναι ταυτόσιμες και τρεις υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τώρα, για το πρώτο τμήμα... Τις 113. Το δεύτερο δεν είναι παραδεκτό. Γιατί δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη ε, πρόταση. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 114 δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 115 δεκαπέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται ε, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα συμβαστική 9 υπέρ κατά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 αποχές ε, ε, απορρίπτονται 152 247 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.48 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίθηκε 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 έλεγχος okay. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Σίγουρα, σαφέστατα εγκρίνεται. Ε, είχα ερμηνεύσει πλημελώς ένα τμήμα. 161 είναι συμβατή με την 160 υπέρ. Κάτα αποχές εγκρίνεται. Συμβασική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα, συμβατική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, unblock 202 και 251 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Avete votato tutti. Il voto è chiuso. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.17 και 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 2.18 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Unblock. 2.19 και 72 υπέρ κατά αποχές α, με εγκρίνονται. 2.31 όχι συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Πράγματι 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 2.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.44 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το τροποποιημένο κείμενο τώρα δια ηλεκτρονικής ψήφου παρακαλώ. Avete votato Έχετε ψηφίσει όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια

Now it is a game, only 30 minutes. Τώρα παιχνιδάκι είναι αυτό, μόνο 30 τροπολογίες έχουμε. Επόμενο σημείο είναι η ψήφος το 30 και 31η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του, της νομοθεσίας η κυρία Γκούτελαντ είναι η συγκήτρια μπορούμε να ξεκινήσουμε τροπολογία 1 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά ελέγχουμε. Avete votato tutti? Πέρας της ψηφοφορίας. Approvato. Εγκρίνεται. 3. Iper. Catà. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 συμβατή με τη συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 συμβατή με την συμβαστική. Υπέρ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 Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία εγκρίθηκε. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Abbiamo adesso l'emendamento 30. Chi ha fatto? 30 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Δεν είμαστε, δεν έχουμε καθυστερήσει. Ίσα ίσα. Πέρα τη πληροφορία. Απορρίπτεται. 29-29. Καλά κάναμε και το ελέγξαμε. 31. Υπέρ κατά αποχές τα ίδια έλεγχος Avete votato tutti? Ψηφίσατε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να ελέγξουμε. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Πέρασε. Ενεγκρίθη. Με πολύ μικρή διαφορά. Λοιπόν, 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου παρακαλώ Avete votato tutti, il voto è chiuso. Peras ενεγκρίθη. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκούτελαντ, η οποία δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει. Συγχαρητήρια της. Okay, we have uh, some... Πέντε λεπτά διακοπή και μετά θα πάμε στην έκθεση για τον προπολογισμό. Dear colleagues, uh, Συνάδελφοι, έχουμε τον κύριο Φερνάντες, που είναι ο γενικός μας ηγητής για τον προϋπολογισμό του 2016 και έχει έρθει για να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω πως είναι μακροσκελέστατη η διαδικασία ε, σύνταξη εκτέλεση του προπολογισμού. Ξέρω γιατί ήμουν και εγώ εισηγητή στο παρελθόν. Και τι κάνει συνήθω ο εισηγητή, Κάνει μια γύρα σε όλε τι επιτροπές και ε, τους μιλάει για τις προτεραιότητες ε, για το επόμενο ε, οικονομικό έτος Επίσης μας εξηγεί τις βασικές δυσκολίες στις οποίες πρέπει να αντεπεξέλθουμε και σίγουρα θα κάτι θα μας πείτε και για τις πληρωμές, έτσι. Είναι ένα ε, σύνθεση πρόβλημα που στις αρχές της διαδικασίας ε, κατάρτιση του προϋπολογισμού χρειάζεται κάθε φορά να λύσουμε. Αλλά να μην πολυλογώ εγώ να δώσω στον κύριο Φερνάντες το λόγο για να αρχίσει μια ώρα αρχίτερα και η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Έρχομαι για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες, αλλά κυρίως για να σας ακούσω. Να υποφεληθώ από τη σοφία σας, να ακούσω τις απόψεις σας και έτσι να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, γνωρίζει εκ των έσω τη διαδικασία, κατέχει τη διαδικασία και ε, υπήρξε και ο ίδιος ηγητής και ξέρει ακριβώ πώς λειτουργεί. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι στην Ολομέλεια της 11ης Μαρτίου 2015 εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές ε, και έχουμε τα τρία ε στα αγγλικά απασχόληση, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλος ιδιαίτερος και επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει αντίκτυπο στις γραμμές του προϋπολογισμού και δεν ξεχνάμε και την εσωτερική αλληλεγγύη και την εξωτερική αλληλεγγύη καθώς και την ασφάλεια και την μετανάστευση. Βασιζόμαστε επί αρχή ότι θα τηρηθούν ε, οι υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, οι συμβασμοί στους οποίους έχουμε καταλήξει και αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Με το Συμβούλιο Καταλήξαμε σε ε, μία συμφωνία. Έχουμε προγραμματίσει τις ε, μη καταβληθήσεις ε, πληρωμές και υπενθυμίζω ότι οι πληρωμές απορρέουν φυσιολογικά από τις αναλήψεις υποχρεώσεων και υπό φυσιολογικέ συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουμε πρόβλημα με τις πληρωμές γιατί έχουμε ήδη αναλάβει τη δέσμευση και δεν μιλάμε για φρέσκο χρήμα, για νέα κονδύλια, μιλάμε για τιμολόγια τα οποία πρέπει να εξοφληθούν προγράμματα που έχουν ήδη εκτελεστεί και για τα οποία έχουν δώσει σύμφωνη γνώμη ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί στην περίοδο 2007-2013 η πολιτική συνοχή, που είναι και το βαρύτερο σε σημασία ζήτημα Έχουμε καταλήξει σε συμβιβασμό για το 2016 να έχουμε κατά το όριο 2 δις ε, μη ε, εκτελεστήσεων πληρωμών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπήρχε συμφωνία για το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή έχουμε δώσει τη σύμφωνη γνώμη τα κράτη-μέλη και μετά διαφωνούν για τον προπολογισμό, ο οποίος έχει καταρτηθεί όμως ε, επί τη βάση του πολιετούς και να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ένα νέο στοιχείο, η ευελιξία, η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα περιθώρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Είναι ο όρος που θέσαμε για να καλύψουμε το ε, κενό που υπήρχε στον προϋπολογισμό ε, και τις περικοπές που έπρεπε να γίνουν παρότι, παρά τη διεύρυνση. Ε, ο προϋπολογισμός 145 δις δεν ξεπερνάει το 1% του ΑΕΠ και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πώς προκύπτει με σαφήνεια ε, η προσθέμενη αξία του προπολογισμού. 6% είναι τα λειτουργικά έξοδα για τη διοίκηση. 94% ε, είναι επενδύσεις από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ε, προφανέστατη απόδειξη της προσθέμενης αξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει σε σχέση με το Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων, επειδή βασιλήκαμε στον Ένωση 2020 και το ΣΕΦ, ένα δις, πήραμε το περιθώριο που δεν ήθελε το Συμβούλιο, ε, το οποίο όμως αποδεικνύει πως θα είναι αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο για να υπάρχει σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ε, τώρα, χρονοδιάγραμμα διαπραγματευτική εντολή για τον Τρίλογο 23 ε, Ιουνίου στην ε, Επιτροπή, 3, ε, εδώ τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Μετά έχουμε τις πρόθεση τροπολογιών πριν το καλοκαιρινή διακοπή, το, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο σε Επιτροπές. 23 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουν οι τροπολογίες τη Επιτροπή Προϋπολογισμών. Μετά το ψήφισμα 23 Οκτωβρίου ψηφίζουμε στην Ολομέλεια και μέχρι τις 18 Νοεμβρίου συνδιαλλαγή. Για τις προτεραιότητες της ΕΜΒΗ βλέπουμε ότι στο ε, τίτλο 2 έχουμε το πρόγραμμα LIFE. Σε... Έχουμε αύξηση 6,4% για την ανάλυση υποχρεώσεων και 1,4% αύξηση για τις πληρωμές. Για τον τίτλο 3, το Food and Feed, για το πρόγραμμα για την υγεία 2,1% αύξηση για την ανάλυση υποχρεώσεων food and feed 4% για την υγεία, πάλι θα ανάλυση υποχρεώσεων και για τις πληρωμές το food and feed 28,6% αύξηση για τις πληρωμές και για την υγεία 23,1%. Αυτές οι αυξήσεις στις πληρωμές αποσκοπούν επίσης τον περιορισμό των, μη, ε, των ανεξόφλητων λογαριασμών στις περισσότερες περιπτώσεις. Για τον ΕΦΣΑ, το ACDC και το EA βλέπετε ότι ε, υπάρχει πρόταση μείωσης 2%. Αυτό σημαίνει πως Ε, σε τα πέντε χρόνια θα είναι 10%, δηλαδή είναι περισσότερο από το 5% που προβλέπεται, η μείωση που προβλέπεται για όλα τα ε, θεσμικά όργανα. Ε, βλέπουμε ότι δεν άλλαξε ο αριθμός των θέσεων για τον ΕΜΑ, για τον ΕΟΦ Ε, και μπορούμε να πούμε και να μπούμε και σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε για κάθε μεμονωμένη περίπτωση έχουμε επίσης για τα πιλωτικά προγράμματα στον τίτλο 3 έχουμε ένα πρόβλημα. Θα εξαντλήσουμε το περιθώριο και μάλιστα η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το όργανο ευελιξίας ε, για 124 εκατομμύρια και ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία για να μπορέσουμε να έχουμε πιλωτικά προγράμματα σε αυτό το τίτλο 3. Τα πιλωτικά προγράμματα, υπενθυμίζω, πως τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις ε, εκτελούνται υπό του δημοσιονομικού κανονισμού 100 εκατομμύρια κατανότατο ρε για τις προπαρασκευαστικές και 40 εκατομμύρια για τα πιλωτικά. Φυσικά, σας το είπα, και το επαναλαμβάνω, ήρθα κυρίως για να σας ακούσω, να με βοηθήσετε, τα φώτα σας να μου δώσετε για να έχουμε τον καλύτερο προϋπολογισμό. Θα σημειώσω τις απόψεις και τις προτάσεις σας. Γι' αυτό και θα σιωπήσω. Ευχαριστούμε, Ζωζέ Μανουέλ. Ξεκινώ αμέσως εγώ δίνοντας τις προτεραιότητες τρόπον την της Επιτροπής καθότι ασχολούμαι με τα θέματα προϋπολογισμού. Σίγουρα κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα ζητήσουν το λόγο και θα συνεισφέρουν ώστε να ενισχύσουμε τις ενδείξεις που θέλει η Επιτροπή αυτή να σου δώσει για τη διαδικασία του προπολογισμού. Είμαστε πλέον στο, στο τρίτο έτος ε, του πολίτους ε, δημοσιονομικού στο οποίο θα έπρεπε κανονικά να κυλούν κανονικά ομαλά τα προγράμματα συχνά ωστόσο καθότι έχουμε κάποιες δυσκολίες με τις πιστώσεις Ακόμα και στο live έχουμε καθυστερήσεις ε, και κενά σχετικά με τις ελλείψεις αυτές. Και ως Επιτροπή σημειώνουμε ότι οι πόροι του νέου έτους για τον προγραμματισμό live θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το πολιετές δημοσιονομικό και όχι κατώτεροι από το προηγούμενο έτος και επομένως θα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα προτεραιότητος για την Επιτροπή μας. Από την άλλη μεριά έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα υπό τον τίτλο 3 και όπως γνωρίζεις υπάρχει μια περιπλοκότητα στο 3 μικρών και πολύ μικρών προγραμμάτων για την Ευρώπη των πολιτών και που προφανώς συνδέονται με τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, των μέσων πολιτικής προστασίας κτλ. Εμείς θα ζητούσαμε και αυτά τα προγράμματα για το προϋπολογισμό του 2016 να έχουν, να τύχουν της απαραίτητης προσοχής και να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την υψηλή χρησιμότητα που έχουν ε, και την ωφέλεια που έχουν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς θα θέλαμε όλα τα κονδύλια προορίζονται στο κλίμα, το περιβάλλον, την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πολύ συχνά είναι περιορισμένα να διατηρηθούν εν πάση περιπτώσει στα προηγούμενα επίπεδα διότι τα θεωρούμε πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες και να σημειώσω και κάτι για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΦΣΑ, ΕΜΑ και διάφορες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου της Επιτροπής αυτής. Και αυτό το θέμα των οργανισμών αυτών είναι σημαντικό γιατί συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι η μείωση του προσωπικού έχει κόστος και δεν είναι δεν συνάδει με τις ανάγκες των οργανισμών οι οποίοι καλύπτονται εξωτερικά για να προβαίνουν σε δραστηριότητα σύμφωνα με την εντολή που τους έχουμε δώσει. Εάν λοιπόν οι εξωτερικοί πόροι υπολογιστούν στον προϋπολογισμό καθότι απαιτούν και τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους, το σχέδιο της μείωσης του προσωπικού κάποιες φορές συχνά δεν ευθυγραμμίζεται προς τις εντολές που έχουμε δώσει στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες αυτές και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Διότι αφενός μπορεί να θέλαμε όσοι νομοθέτες να προχωρούν σε περισσότερες δραστηριότητες και να αντλούν τους πόρους από την αγορά δεν μπορούμε να το ζητούμε να μειώνουν το, το προσωπικό διότι δεν θα μπορούσαν πλέον να ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Αυτά είναι που θέλουμε να σου διαβιβάσουμε ως Επιτροπή και θέλουμε αυτό να συμπεριληφθεί στη διαδικασία και στη διαπραγμάτευση που σίγουρα θα είναι δύσκολη αυτή που θα κάνεις στο τέλος με το Συμβούλιο Τώρα εδώ θα έδινα το λόγο σε όποιον συνάδελφο τον θέλει. Κροστέτε, γκρότε, μετά βλέπουμε. Φρονσουά, τέλος πάντων. Ναι, πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω το συνάδελφο για την πολύ δύσκολη δουλειά και την πολύ δουλειά γνωρίζουμε Ήθελα να στηρίξω απολύτως τα όσα σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ιδιαίτερα για τα θέματα υγείας. Επομένως, συμφωνώ απολύτως για τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες που μας αφορούν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Συνέχεια του ζητούμε περισσότερα και κάποια στιγμή έρχεται δηλαδή η στιγμή που δεν μπορούν πλέον να κάνουν τη δουλειά που τους ζητούμε. Εφόσον δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Άρα, Υπάρχουν οργανισμοί που είναι υπερβολικά σοβαροί, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δεν μπορεί να προβλέπουμε για τέτοιους οργανισμούς να προβλέπουμε μειώσεις προσωπικού. Για τα θέματα πάντοτε υγείας που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πόροι που αφαιρούν άμεσα και στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Ερεύνης, εξάλλου διότι υπάρχουν θέματα που άπτονται και της έρευνας και της ε, πολιτικής ε, υγείας και είναι απολύτως απαραίτητο εκεί να εγγραφούν τα όσα πρέπει να εγγραφούν. Διότι ε, και ακόμα εντός της εβδομάδας γίνονται συζητήσεις σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του κανονισμού για τα παιδιατρικά, για τα ορφανά παιδιά, για τα κοινοτόμα φάρμακα. Υπάρχουν ένα ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια αυτά γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην έρευνα. Και κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι η Κομισιόν δεν δίδει επαρκή προσοχή σε αυτά τα θέματα υγείας στο γενικό προϋπολογισμό και επομένως εμείς πρέπει να καταδείξουμε τη βούλησή μας για θέματα που έχουν άμεση σχέση, άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες και μια αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. ich möchte auch noch mal ε, Γκρότε, το ίδιο θέλω να πω κι εγώ και να τονίσω και πάλι ότι οι εξωτερικοί αυτοί οργανισμοί έχουν και πελάτες. Ε, ε, εμείς αν μειώνουμε το κόστος και ε, οι πελάτες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και αυξάνονται και οι προθεσμίες και οι χρόνοι αναμονής είναι άδικο. Εγώ είμαι ο σύνδεσμος για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έμα. Ε, θα πρέπει να δίνονται οι αδειοδοτήσει και οι εγκρίσει σχετικά σύντομα. Δεν μπορεί να τους αφήνει να περιμένουν και να τους βάλει ένα τέτοιο στενό κορσέ που το κάνει η ίδια η Επιτροπή για τον εαυτό τη. Και κάνει και τεχνάσματα. και με ταχυδαξιλουργίες δείχνει ότι μειώνει το κόστος και το προσωπικό ε, και ε, για την Επιτροπή μας και ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πελάτες ε, που πρέπει να εξυπηρετούνται σε ένα λελογισμένο χρονικό διάστημα και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό γίνεται μόνο όταν στις περιόδους αχμής υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό και θα πρέπει να είναι ευέλικτη η κατάσταση. Γιατί όταν δημιουργείται από ένα κανονισμό ή από μια ε, νομοθεσία, ένας τέτοιος οργανισμός έχει και ένα ρόλο ε, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαφορετικά αυτά τα χαρτιά στη θεωρία αλλά όχι στην πράξη. Οι οργανισμοί αυτοί εξωτερικοί θέλουν αέρα να αναπνεύσουν, δεν μπορούμε να τους τραγκαλίζουμε. Τα είπε και η Φρανσόας Γκροστέτ και νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή μας να τους δίνουμε αυτό το περιθώριο, αυτή την ανάσα. Γιατί αυτόνομη είναι έτσι κι ε, θα πρέπει να βρούμε δρόμους ε, πρακτικούς και εφαρμόσιμους. Ο Γιάνν Γκερμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φερνάντες για την παρουσία του. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι για τους εξωτερικούς οργανισμούς, αλλά έχω διαφορετική άποψη που θέλω να καταθέσω. Εμείς εστιάζουμε περισσότερο στις επιδόσεις του προϋπολογισμού. Ε, δηλαδή, πιστεύω ότι όλη η διαδικασία του προπολογισμού παρά είναι τεχνική, έτσι δεν είναι. Κάθε φορά ξανά και ξανά αυτή την τεχνοκρατική άσκηση. Εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Spend. Θέλουμε αποτέλεσμα από τα χρήματα που δαπανούμε. Ας πούμε για το περιβάλλον έχουμε το LIFE 3,4 δις για το περιβάλλον σε αυτό το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την προγραμματική περίοδο με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και από την άλλη έχουμε ένα τμήμα της γεωργικής πολιτικής που λέγεται το αγροπεριβαλλοντικό ε, σύστημα που είναι 22 εκατομμύρια για την επταετία αυτή, δηλαδή 7 φορές λιγότερο. Αλλά οι επιδόσεις, τα αποτελέσματα των 22... Ε, δισεκατομμυρίων δεν μπορούν να μετρηθούν. Το ελεκτικό συνέδριο δεν βρίσκει που πήγαν αυτά τα 22 δις που είναι για το περιβάλλον στη Γεωργία. Και εδώ πιστεύω ότι έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Το πρόγραμμα Live είναι πάρα πολύ επιτυχές. Ε, η θέση του προπολογισμού που πάντα ε, ε, λείπουν χρήματα. Και στη γεωργία τα περιβαλλοντικά έχουμε επταπλάσιο, αναλαμβάνω ποσό, χωρίς αποτέλεσμα. Είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο έχει τονιστεί και από το ελεκτικό συνέδριο. Και θέλω να παραθέσω μια παράγραφο ε, στην ετήσια έκθεση του 2013 όπου λέγει το Ελεκτικό συνέδριο έχει διαπιστώσει ότι η επιλογή προγραμμάτων ε, εστιάζεται κυρίως ε, στο να απορροφηθούν κονδύλια που αλλιώ θα χαθούν ε, και αυτό, αυτή είναι η πρώτη τους σκέψη. Η δεύτερη να δουν εάν ε, τηρούνται οι κανόνες και σε περιορισμένο μονοβαθμό και τρίτο κριτήριο είναι η επίδοση. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας να πιάνουν τόπο ως πολιτικοί, να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι ο ευρωπαϊκός υπολογισμός έχει τεράστια προστιθέμενη αξία ότι παράγει υπεραξία και δεν τον έχουμε τον προπολογισμό αυτόν τον ευρωπαϊκό μόνο για να ξοδεύουμε χρήματα. Δεδομένων λοιπόν αυτών των συμπερασμάτων του ελεκτικού συνεδρίου και του παραδείγματος που σας έδωσα για το προϋπολογισμό live από τη μια και τα άλλα τα περιβαλλοντικά της γεωργίας, είστε διατεθειμένος να εστιάσετε πολύ περισσότερο λοιπόν στα αποτελέσματα και στα πεπραγμένα του προϋπολογισμού του 2016. Ευχαριστώ κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Φερνάντη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μας ενημερώσετε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Επανέρχομαι ε, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Την ε, το περασμένο έτος είχαμε προβλήματα με το έμπολα. Και είχαμε το στρατηγικό έγγραφο, ε, έγινε δουλειά για τον συντονισμό και τις διαδικασίες. Σήμερα έχουμε λιγότερους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την επαγγελματικότητα και την αριστεία αυτής της δουλειάς, πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα κονδύλια. Εφόσον θεωρούμε δηλαδή ότι χρειαζόμαστε τον οργανισμό αυτόν. Και από ό,τι φαίνεται τον χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε χωρίς προϋπολογισμό. Η θα είναι ένα κενό γράμμα και δεν θα βοηθάει σε τίποτα. Επίσης έχουμε υψηλές ε, προκλήσεις ε, και προβλήματα από διάφορες ε, νόσους, φυματίωση, πατήτιδα κτλ. και όπως είχε αναφέρει και ο συνάδελφος Δεκορέα. Τι θα κάνουμε με όλα αυτά εφόσον ο οργανισμός δεν έχει επαρκείς πόρους. Εγώ δεν έχω απάντηση. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ για μία ακόμα φορά να περικοπεί ο προϋπολογισμός του οργανισμού. Διότι θα δημιουργήσουμε μια πολύ προβληματική κατάσταση που τελικά θα επιφέρει πολύ ψηλότερο κόστος από αυτό που εξετάζουμε ως περικοπή. Στην Επιτροπή προεπολογισμού εξετάζουμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ή στην ε, δημιουργία μιας καινούριας έδρας. Και εξερευνούμε ακριβώς και τις όποιες δημοσιονομικές ε, δυνατότητες έχουμε. Εγώ διαμαρτύρομαι για τις περικοπές αυτές προϋπολογισμού και για αυτόν τον οργανισμό και για τις προηγούμενες όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι. Και κάθε χρόνο τα ίδια λέμε ότι είναι πολύ σημαντικοί οργανισμοί, ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς, ότι είναι αξιόπιστοι, ότι τους χρειαζόμαστε και συνεχίζουμε να περικόπτουμε τον προπολογισμό. Δεν είναι συνεπή όλα αυτά. Ευχαριστώ, λέει κύριε Ζαβόρ. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να μας μιλήσετε για το προϋπολογισμό του 16. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις ε, βασικούς ε, τομείς. Όπως είπε ο κύριος Γκεμπράντη, Μιλάμε για τις γραμμές του προϋπολογισμού που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, έχουμε υπόψη τις δραστηριότητες και τις πολιτικές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ε, υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Επιτροπής ΕΜΒΗ, επηρεάζουν όμως σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον. Σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού θα πρέπει να φροντίσουμε δεν υπάρχουν δαπάνες που να αντιβαίνουν στις προσπάθειες που κάνουμε με τις δικές μας γραμμές του προϋπολογισμού. Δεύτερον, πολύ σημαντικό σημείο, η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Το live τον έφεραν οι συνάδελφοι, πέραν αυτού Υπάρχει το Natura 2000, ε, το δίκτυο που έχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μεγάλο αριθμό των κρατών μελών διαπιστώνεται πρόβλημα χρηματοδότησης σοβαρό για το δίκτυο Natura 2000. Έχοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ε, και τη δέσμευση να την αναθεώρηση των οδηγιών για τα πουλιά και τους βιοτόπους που είναι τα δύο ερίσματα ουσιαστικά του Natura 2000 θα πρέπει να ε, φροντίσουμε ώστε να υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση και σωστή εκταμίευση προτού αρχίσουμε με τις εργασίες της αναθεώρησης ε, των ε, ισχυρών κανονισμών τρίτη και τελευταία παρατήρηση οι οργανισμοί. Θα συμφωνήσω πολύ με τους συναδέλφους μου. Ήθελα μόνο να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, ΕΦΣΑ, με το νέο κανονισμό για τα ε, μεταλλαγμένα που θα αρχίσει να ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι θα αυξηθεί πάρα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο φόρτος εργασίας της ΕΦΣΑ και θα έχουμε ε, αιτήσει για εγκρίσει ε, για νέου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και εφόσον αναμένεται αύξηση του έργου του, της ΕΦΣΕ είναι ανεύθυνο νομίζω να ε, περικοπεί ο προπολογισμό του οργανισμού, διότι ενδέχεται αυτό να οδηγήσει σε περιβαλλοντικούς κινδύνους που θα προκληθούν από γενετικά τροποποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φυσικά ε, απέφχεται ο λαός της, ε, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω αυτά ε, που είπαν οι προλαλήσαντες. Αυτό που μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ίδια και ορίζονται και από τις συνθήκες αυτό. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα ε, στο άρθρο 168 από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρόκειται για όλα τα θέματα που άπτονται της υγείας και όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ε, διατηρούν και να αναπτύσσουν το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του Ευρωπαίου πολίτη. Και αυτό γίνεται μόνο με τους αντίστοιχους οργανισμούς και θα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά στην πράξη. Η απέτηση λοιπόν για ε, καλύτερη δυνατότητα λειτουργίας για περισσότερους πόρους και οικονομικούς για τους οργανισμούς είναι προϋπόθεση και προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καν στο άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Φερνάντες, θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλούμε για το σχέδιο προεπιλογισμού της ε, Κομισιόν και ότι το Συμβούλιο θα έχει ανάγνωση του σχεδίου αυτού. Και κανονικά θα έχουμε άσχημα νέα από το Συμβούλιο. Κανονικά συμφωνώ με τα όσα ελέγχθησαν, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πόσο κοστίζουν αυτά που περικόπτουμε. Πόσο κοστίζουν οι εξοικονομήσεις δηλαδή. Γιατί όταν θέλουμε αποτελέσματα από τους οργανισμούς είναι, υπάρχει ένα εκατότατο όριο υπό του οποίου δεν μπορεί πλέον ο οργανισμός να ανταποκριθεί. Και αυτό δεν είναι καλό για την ανακοίνωση και πρέπει να το σκεφτούμε. Για τα θέματα εφαρμογής και αποτελεσματικότητας βεβαίως και είμαστε υπέρ της πειθαρχία και της σοβαρότητας. Βεβαίως και είμαστε σε ένα πολιετές δημοσιονομικό με καινούριε πολιτικές ε, συνοχής όπου το περιβάλλον είναι παρόν με νέα πολιτική συνοχής στην οποία την οποία μάλλον πολλές χώρες χρησιμοποιούν για τη μεγέθυνση αλλά και για την ε, έρευνα και την καινοτομία. Επομένως τα θέματα της, των επιδόσεων ή της αποτελεσματικότητας είναι κάτι που θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Όπως και τα όποια αποτελέσματα. Τι προσπαθώ να πω. Εάν δεν έχουμε, δεν προχωρήσουμε σε διαγωνισμό εντός ε, προγράμματος, στο τέλος θα πούμε ότι δεν, υπήρχε, δεν υπήρξε εκτέλεση και άρα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Πρέπει να βλέπουμε και τους λόγους δηλαδή της μη εκτέλεσης. Αν δεν προχωρούμε σε διαγωνισμό πώς να εκτελεστεί. Αν κινούμαστε με καθυστέρηση στα επιχειρησιακά των χωρών, προφανώς και θα έχουμε χαμηλότερη εκτέλεση. Έχουμε νέα πολιτική συνοχή όπως έλεγα, αλλά έχουμε και νέα γεωργική πολιτική. Για το life συμφωνώ απολύτω. Και μάλιστα έχω ανάγκη από τη στήριξή σας για τις διαπραγματεύσει. Θυμίζω ότι η θέση του Συμβουλίου θα είναι ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρός, το Συμβούλιο θα προσπαθεί σε κάθε ανάγνωση να τον κάνει ακόμα μικρότερο και με κάθε νέα θέση του θα προσπαθεί να μην αναλαμβάνει περαιτέρω δεσμεύσεις. Δηλαδή υπάρχουν και τα άλλα θεσμικά όργανα και όχι μόνο το Κοινοβούλιο. Σημειώνω πάρα πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις και ήδη βρίσκονται στην μεγάλη τους πλειοψηφία στην έκθεση. Και βεβαίως το θέμα των οργανισμών θα είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο στη διαχείρισή του. Και ελπίζω, ελπίζω, εύχομαι να έχουμε μια ανάγνωση του Συμβουλίου που να μην οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα προβλήματα γιατί ήδη αρκετά έχουμε με το σχέδιο της Κομισιόν. Αλλά θα περιμένουμε την ανάγνωση και θα συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή για να προσπαθήσουμε να έχουμε και τις δικές σας, να καλύψουμε μάλλον και τις δικές σας ανησυχίες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε και αρνητικές προτεραιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε φτάνουμε πλέον σε μια άλλη συζήτηση για μια άλλη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ζωζε Μανουέλ. Ευχαριστούμε που έλαβα υπόψη σου τις ε, προτεραιότητες μας. Και θέλουμε να τονίσουμε εκ νέου ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους οργανισμούς. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη το αίτημα της Επιτροπής αυτής. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συναδέλφους και εσένα προσωπικά για τη ζήτηση αυτή. Για το χρονοδιάγραμμα έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης 15 ή 16 Ιουλίου το κορεπέρ που θα εγκρίνει θέση Συμβουλίου μέσα ή τέλη Ιουλίου και προθεσμία τροπολογιών για την Επιτροπή αυτή θα είναι 17 Ιουλίου. Εδώ μπορούμε να κλείσουμε, πιστεύω, το πρωινό και θα δούμε τι θα γίνει το απόγευμα. Καλή σας όρεξη.